Ε, το νερό. Έχουμε συγκεντρώσει και υπογραφές με ένα δημόσιο δημοψήφισμα κατά το ιδιωτικοποίηση του νερού της διανομής του νερού και συγκεντρώνουμε ακόμα τέτοιες υπογραφές σε μεγάλο αριθμό. Συνάδελφοι, μόλις έλαβα την πληροφορία πως θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση όσον αφορά τον αντιπροέδρο, την άφηξη του αντιπροέδρου Biden. 10-15 λεπτά καθυστέρηση, οπότε συνεχίζουμε με την επεξήγηση των ψηφών. Πριν το κάνω αυτό, να έχω και μια άλλη ανακοίνωση. Να καλωσορίσω μια μαροκινή αντιπροσωπεία Να τους ενημερώσω κιόλας ότι στο πλαίσιο των ε, διακοινοβουλευτικών επαφών αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ μια μαροκινή αντιπροσωπεία. Μαροκινοί βουλευτές βρίσκονται εδώ σε επίσκεψη εργασίας. Στο πλαίσιο της επαφής ε, της ε, Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μαρόκο. Συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Μαροκινού Κοινοβουλίου και ο κ. Παντσέρη, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαπιστώνει με ικανοποίηση πω οι σχέσει μεταξύ τη Ένωση και του Μαρόκου είναι εξαιρετικέ. Και επίσης έχει εγκριθεί το κείμενο που δίνει στο Μαρόκο ε, ιδιαίτερο καθεστώς ώστε να γίνουν διαπραγματεύσεις σε μεγαλύτερη έκταση για κοινά θέματα ενδιαφέροντος. Ελπίζω πως οι συναντήσεις σας ήταν καρποφόρες και έτσι η σχέση μεταξύ των δύο κοινοβουλίων μας θα γίνει ακόμα καλύτερη. Επόμενο σημείο στις επεξηγήσεις ψήφων Απαγόρευση δηλαδή τεχνολογιών που χρησιμοποιούν και ανούχα άλατα για την εξόριξη μετάλλων. Εδώ έχουμε τον κύριο Μεσάρος που θέλει να κάνει επεξήγηση ψήφου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να επεκταθεί η απαγόρευση